Herr Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen. Επαναρχίζουμε τη συνεδρίασή μα. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην ημερήσια διάταξη. Εάν όχι, έχουμε εγκρίνει τα πρακτικά. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης που είναι η συζήτηση για κατεπήγοντα θέματα, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Ξεκινάμε με το θέμα κατάσταση των ακτιβισμών των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη και το Λάος.